Okay. May I ask Καλησπέρα. Καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Ω ήθιστε αρχίζουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. εγκρίνεται. Στη συνέχεια, ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων έχει λάβει 8 σχέδια με, διορθώσεις, με διορθώσεις. Πρόκειται για τα καλυμμένα ομόλογα, πρόκειται τα καλυμμένα ομόλογα και την εποπτεία. Πρόκειται για την προληπτική εποπτεία επενδυτικών εταιριών ε, και τροποποιητικών οδηγιών 2013-36-2014-65. Πρόκειται για τις απαιτήσει του προληπτικού ελέγχου επενδυτικών εταιριών. Πρόκειται για την ε, βιωσιμότητα ε, στον ε, δημοσιονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Πρόκειται για το κλίμα και τα κριτήρια όσον αφορά την κλιματική μετάβαση. Πρόκειται για την πρόθεση των αγορών όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αναπτυξή τους. Πρόκειται για το ΕΜΗΡ 2.2 τις απαιτήσει για την αναγνώριση τρίτων χωρών έχουν κυκλοφορήσει τα σχέδια των διορθώσεων αυτών στους ευρωβουλευτές μέλη της ΕΚΟΝ στις 3 και 4 Οκτωβρίου σε όλες τις γλώσσες. Σύμφωνα τώρα με το άρθρο 241 του κανονισμού, εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ενστάσεις από την Επιτροπή μας, τα διορθωτικά αυτά θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ανακοινωθούν στην πρώτη ολομέλεια του Οκτωβρίου και θα εγκριθούν εκτός εάν υπάρχει αίτημα από πολιτική ομάδα ή από ευρωβουλευτές, 38 ευρωβουλευτές, που θέλουν να τεθεί σε ψηφοφορία το σύνολο των διορθωτικών αυτών. Αυτή ήταν η μία ανακοίνωση. Δεύτερη ανακοίνωση. Θέλω να ενημερώσω τους ευρωβουλευτές ότι δεν θα συνεδριάσουμε τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου. Επόμενο θέμα. Πρόκειται για το σχέδιο έκθεσης που έχουμε όσον αφορά την εξαποστάσεως πώληση αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών. Ο εισηγητής μας είναι ο Ντρέι Κοβάρικ από την ομάδα Renew. Έχουμε και τους ε, σκιώδεις ε, από το ΕΛΚ πρώτα απ' όλα, Γιώργο από το Σοσιαλιστές, μόλις κάτω ε, από τους Πράσινους, και η Α, ναι, λέει ο Και ο Κουσμάου Γκούε, που δεν τον βλέπω εδώ ακόμα. Λοιπόν, το λόγο στον εισηγητή για τις αγωγικές παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή μας και τους σκιώδες εισηγητές για τη δυνατότητα που έχουμε να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά αυτό το θέμα σήμερα. Από ό,τι θα καταλάβετε, με αυτά που θα σας πω σε λίγο, επήγει να προχωρήσει ο φάκελος αυτός και ελπίζω να τα καταφέρουμε σήμερα πρόταση για την ως πώληση αγαθών και ορισμένες εγχώρες παραδόσεις αγαθών προβλέπει μέτρα για ένα καθεστώς ΦΠΑ που θα αρχίσει να ισχύει το 2021. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει διάφορε τροπολογίε όσον αφορά την ως πώληση αγαθών και ορισμένε χώρε παραδόσει αγαθών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι υπάρχουν λεπτομερεί κανόνε που επιτρέπουν την ε, πλήρη λειτουργία ε, των νέων κανόνων όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα αρχίσουν να ισχύουν μέρος του πακέτου που έχει να κάνει με το τελικό καθεστώς ΦΠΑ. Το Συμβούλιο κατέληξε ήδη σε μια προσέγγιση τον Μάρτιο που μας πέρασε και η προσέγγιση του Συμβουλίου και οι τροπολογίες ε, του Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι τώρα ευθυγραμμιζόμαστε ε, γενικότερα με τους κανόνες ε, ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα καλείται να γνωμοδοτήσει επί τη προτάσεω αυτή, ε, προηγουμένω εγκρίνει τι τροποποίησει αυτέ στο Συμβούλιο. Όσον αφορά λοιπόν τη διαδικασία τώρα και τι ισχύει στην Επιτροπή μα, πρώτα είχαμε διαβούλευση συνάντηση με του συντονιστέ και με του σκιώδει εισηγητέ από τι διάφορε πολιτικέ ομάδε και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε με απλοποιημένη διαδικασία η άποψή μα είναι να στηρίξουμε τις τροπολογίες του Συμβουλίου στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι ετοιμάσαμε ανάλογα και ε, την δικιά μας τη γνωμοδότηση. Προκειμένου να λειτουργήσουν πράγματι οι νέοι κανόνες πλήρως από το 2021, ο χρόνος πιέζει. Πρέπει δηλαδή οι δικές μας διαδικασίες να προχωρήσουν γρήγορα. Εξού και οι συντονιστές προτείνουν να ακολουθήσουμε την απλοποιημένη διαδικασία. Έτσι θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία και να επιτρέψουμε τις χώρες μέλη να ξεκινήσουν να ενσωματώνουν τους νέους κανόνες στην εθνική τους ε, νομοθεσία έγκαιρα ώστε να μπορέσει το ηλεκτρονικό εμπόριο να αρχίσει να λειτουργεί πραγματικά από το 2021. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, τώρα Ελκ, παρακαλώ. Ήθελα να ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο Κόβαρη και αυτή την πολύ καλή συνεργασία. Συμφωνούμε με την απλουστευμένη διαδικασία και υποστηρίζουμε τις ε, τροπολογίες. Είμαι πεπισμένος ότι όλη αυτή η πρόθεση ε, για να τροποποιηθεί η οδηγία είναι να περιστεί η απάτη στα θέματα του ΦΠΑ, κυρίω για να προστατευτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και οι επιχειρήσεις αυτές να παραμείνουν και στο μέλλον ανταγωνιστικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Ντόλεσσαλ, Κρόνες Φερνάντες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο σκιοδησηγητής μας ε, δυστυχώς ε, δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θα διαβάσω τη δήλωση του εκ του. Εκ μέρους του. Αναφέρει λοιπόν ότι με αυτή την απλούστευμένη διαδικασία ο στόχος μας είναι να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρμογή των κανόνων για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ε, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο κατ' ουσίαν δυστυχεί σε πάνω από 5 δις ευρώ με τους νέους κανόνες, ε, οι online αγορές ε, και αυτές δυστυχώς πρέπει να αντιμετωπιστούν γιατί συμμετέχουν σε αυτή την φοροαπάτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο της έκθεσης, για αυτό που πριν την απλουστευμένη διαδικασία που και εμείς στηρίζουμε και με πολύ μεγάλη μας χαρά να προχωρήσει το θέμα γρήγορα. Ε, το Συμβούλιο έχει τοποθετηθεί το Μάρτιο και τώρα πλέον απόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί. Εμείς λοιπόν στηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ε, θα επιτρέψει να γίνεται καλύτερη αντιμετώπιση των ε, online αγορών. Απλουστεύονται οι αγορές, αγορές για το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ηλεκτρονικές αγορές και αυτές θα πρέπει να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγή, Οι φορολογικέ αρχές θα μπορούν να σχεδώσουν πληροφορίε για τους πελάτες. Όσον αφορά τις, ε, τη φοραπάτη ε, σε σχέση με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μιλάμε για πάνω από 5 δις ευρώ, 7 δις θα είναι μέχρι το 2020. Εμείς στηρίζουμε την πρόταση που ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να κλείσει αυτό το κενό. Πολύ ωραία. Ο κύριος Ιουτζέν Ιουρζίγκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή Οντρέι Κόβαρικ για την γρήγορη και ε, καλή δουλειά που έχει κάνει πάνω στο θέμα αυτό. Όπως αναφέρθηκε, ήταν σημαντικό το Κοινοβούλιο να ενεργήσει γρήγορα, διότι ε, η δέσμη μέτρων για το ΦΠΑ θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021. Γι' αυτό ήταν επιθυμητό να εγκρίνουμε το, ε, την πρόταση αυτή με την απλοποιημένη διαδικασία. Ελπίζουμε ότι έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσουν τη γραφειοκρατία, καθώς ε, και τις ε, αρχές να κλείσουν κάποια από τα νομικά παραθυράκια που υπάρχουν. Γι' αυτό στηρίζω την πρόταση του εισηγητή και επικροτώ το ότι υπάρχει γενική συμφωνία για έγκριση της έκθεσης αυτής. Σας ευχαριστώ κύριε Γιουρζίκα. Δεν βλέπω τον Χωσέ Κουσμάου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μου φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία όσον αφορά την απλουστευμένη διαδικασία. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι υπάρχει προθεσμία για τις αντιρρήσεις 18 Οκτωβρίου Παρασκευή και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα επιβεβαιωθεί, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα θα είναι η πρώτη Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Υπάρχει κάποιο θέμα στα διάφορα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, σύντομα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές ε, για την πολύ επικοδομητική τους στάση. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε έτσι να επιταχύνουμε την υιοθέτηση αυτής ε, της νομοθετικής πράξης και να έχουμε έτσι ε, κανόνες ΦΠΑ κατάλληλους ε, και σύγχρονους. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλα θέματα, θα ήθελα απλά να σας αναφέρω ότι η επόμενη συνεδρίαση πιθανότατα να πραγματοποιηθεί 5η 17 Οκτωβρίου. Θα επιβεβαιωθεί όμως η ημερομηνία, οπότε θα λάβετε σχετικό email. Αυτά λοιπόν, λήξη της συνεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ.